Wir kommen nun zur Abstimmung. Die Ernennung von Sir Julian King. Προχωρούμε στην ψηφοφορία λοιπόν για τον διορισμό του κυρίου Julian King ως επιτρόπου. Είναι μυστική η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben. Ψήφισαν όλοι οι βουλευτές. Ξαναρωτώ, ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Παρακαλώ, βιαστείτε, βιαστείτε κυρία συνάδελφο. Τελευταία φορά ψήφισαν όλοι οι βουλευτές πέρας της ψηφοφορίας. Εψήφισαν 638 βουλευτές, 394 ναι, 161 όχι, 83 αποχές. Διαπιστώρατε λοιπόν η έγκριση του κυρίου Τζούλιαν Κίνγκ ως νέου επιτρόπου. Äh, Και σας συγχαίρω, κύριε Επίτροπε, για την εκλογή σας. Δεν είναι υπερβολή να πει κανεί ότι αναλαμβάνεται καθήκοντα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Και καθώς ήσασταν και από τους περμάχου τη παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι λογικό να αναλάβετε έστω και σε αυτό το στάδιο την θέση του Επιτρόπου. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν αρέσει εδώ, δεν είστε υποχρεωμένοι να μένετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Wir Προχωρώ στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ. Πώ είστε, πώ λέγεται, α, Μάρτι. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με προσοχή άκουσα τα λόγια σας. Και εξηγήσατε στους βουλευτές ότι αν δεν τους αρέσει αυτή η απόφαση μπορούν να αποχωρήσουν από το ημικύκλιο. Θα υπενθυμίσω, κύριε Πρόεδρε, επί του κανονισμού, ότι δεν μας διόρισε ο κύριος Σούλτς, μας εξέλεξε δημοκρατικά ο γαλλικός λαός. Περνούμε στις ψηφοφορίες για, το για την κοινή πρόταση ψηφίσματος για τις Φιλιππίνες δυνάμει του άρθρου 4 παρακαλώ υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 3 τροπολογία 3 υπέρ κατά απόχες επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία παρακαλώ. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλά, επαληθεύουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 2. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται ε, τροπολογία 5 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε στο σύνολό του παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση ψηφίσματος 6 ομάδων για την κατάσταση στην Σομαλία Υπαριθμόν 1 τροπολογία παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πρόταση ψηφίσματος 7 ομάδων για την κατάσταση της Ζιμπάμπουε τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε λοιπόν ηλεκτρονικά πέρα της ψηφοφορίας ε, αρκετή ψηφοφορία, συγγνώμη. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται το, η τροποποιημένη πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό τη υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται και σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε τώρα τις ψηφοφορίες. Έχουμε το πρώτο θέμα. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Ταξιδιωτικό έγγραφο κτλ. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 3. Α2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 33 CP επί της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 34 μπι υπέρ κατά αποχές απερίφθη 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 CP λέει η Πρόεδρος. I can't hear. Check. don't understand. Yeah, no Polish interpretation. No Polish interpretation. There is no Polish interpretation. Just. Μια στιγμούλα γιατί δεν υπάρχει η διερμηνία στα πολωνικά. Ε, τα μικρόφωνα όμως δεν είναι αναμένα για να υπάρξει διερμηνία. Okay, we will continue and... Θα συνεχίσω λοιπόν και θα δούμε πώς πάει. 33 CP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα ονομαστικά παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Και εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια. Τώρα περνάμε στην έκθεση Γέσεκα. Block vote, τροπολογίες επιτροπής υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνονται. Τροπολογίο 1 CP, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2 παράγραφος 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 CP. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 CP. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 CP υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 CP υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε παρακαλώ. The vote Εγκρίνεται. Ναι, αλλά να σηκώνετε και κανένα. χέρι. Πρωτότυπο τώρα, κείμενο, προφορική τροπολογία, ο κύριος Ούρτα Σουν. Ναι, ευχαριστώ. Μία προφορική τροπολογία 36.2 μετά το ΣΥΝΑ λέει δεκατότατες διοικητικές οικονομικές κυρώσεις πρόστιμα τουλάχιστον ίσως με το ε, ποσό των ε, διαφυγών των, ε, μάλλον των κερδών ή των απολειών σε τρίτα μέλη λόγω της παράβασης όταν αυτά μπορούν να οριστούν. more 40. Υπερβαίνουν 40. Δεν γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία. Πηγαίνουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 CP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η πρόταση της τροπής ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Θέλω να ζητήσω αναβολή της ψηφοφορίας ε, με βάση τον κανόνα 61.2 για το νομοθετικό ψήφισμα. Θέτω την πρόταση σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επομένως. Παραπέμπεται στην Επιτροπή το ζήτημα για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Then we go to Πηγαίνουμε στην έκθεση της κυρίας Κέλλερ. Καταρχάς έχουμε όλες τις τροπολογίες άμας επιτροπής ψήφι υπέρ. Block vote. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Όμως, πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας. πρόταση της Κομισιόν. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Report by Mrs. amendment. Τροπολογία Ατζέα. Block vote, τροπολογία επιτροπής. Ψήφι περ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is... Πέρας. Της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. βασικοί objectives για το ΣΥΤΕΣ. η βασική στόχη περ, κατά, ποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Φέρμπερ τώρα. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα το ψήφισμα συνολικά με ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Κάρας. Παράγραφος 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 33 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 35 παράγραφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 39 περ... κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 43, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα, έκθεση Κρασνοντεύσκη, παράγραφος 17. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά πάλι, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, λέει πρόεδρος. Α, συγγνώμη. Τρίτο τμήμα, ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Προφορική τροπολογία. Παρακαλώ κύριε Σιγητά. Uh, like to... Ναι, θα θέλαμε να αλλάξει διατύπωση. Όταν μιλάμε για πρόσθετα διοικητικά βάρη, να λέμε αχρίαστα, unnecessary διοικητικά βάρη. Πρόεδρος, υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία. Όχι. Επομένως, θέτω την ούτως σε παράγραφο σε δύο τμήματα σε ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 31. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ψήφι περ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παράδοση 68 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι ΠΕΡ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. The vote is... Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 74 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 79 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ Against. κατά αποχές εγκρίνεται 80. παράγραφος 80 πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται και δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά The vote is... τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται Αιτιολογική σκέψη Κ, τροπολογία 1. Παρακαλώ ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Π. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Αιτιολογική σκέψη ΤΑΦ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, αιτιολογική σκέψη Υ, ε, ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. αιτιολογική σκέψη το σύνολο του ψηφίσματο τώρα με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στην ε, ψηφοφορία της έκθεσης Weber, παράγραφος 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 2. Σε δύο τμήματα και πάλι. Το πρώτο με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. Παράγραφος 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 35. Ποιος είναι... Σε δύο τμήματα ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 53. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 59. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 παράγραφος. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 68. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 69 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό παράγραφος 77 σε δύο τμήματα Πιο Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 83. Σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην αιτιολογική αναφορά 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη γιου με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία την, ε, της έκθεσης της κυρίας Χάρκιν. Παράγραφος 13 με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 33. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 53. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη Q. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Και αιτιολογική σκέψη R. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Uh, θα συνεχίσουμε. It's time for explanation. Ήρθε η ώρα της επεξηγήσεως ψήφων. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον Χάναν Ντάνιελ.